Ε, λειτουργήμα ή επάγγελμα που είναι συμβίβαστο με την ιδιότητα του Ευρωβουλευτού. Ο πρόεδρος ε, των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών με ενημέρωσε ότι ο κύριος Έντουαρτ Μακμίλαν Σκοτ δεν είναι πια μέλος της ομάδας τους από τις 20 Ιουλίου του 2009. Έλαβα από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και των ε, ε, Ευρωπαίων Δημοκρατών καθώς και των Πρασίνων ε, της Ευρώπης για την Ευρώπη των Πολιτών μερικές, μερικά ψηφίσματα σε σχέση με αλλαγές σε κοινοβουλευτικές επιτροπές και διακοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες τα οποία θα επισυναφθούν στα σημερινά πρακτικά. Αν δεν υποβληθούν παρατηρήσεις ή για τις αλλαγές αυτές θα θεωρηθούν ως εγκεκριμένες.